Liebe Kollegen, wir setzen die Sitzung fort. Ähm, ich äh, begrüße Sie. Es sieht nicht so aus, als wären es viele, aber... Αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται σαν να μην είμαστε πολλοί μέσα στην αίθουσα, αλλά πολλοί είμαστε, απλώς είμαστε έτσι διασκορπισμένοι. Ελπίζω να μπορείτε όλοι να με ακούσετε. Καλωσορίζω τον Υπουργό Παιδείας, εκπαίδευση από την Ισπανία. Είχαμε την τιμή στην αρχή της Ισπανικής Προεδρίας να μιλήσουμε με τον ε, Υπουργό. Χαιρόμαστε που είναι και πάλι εδώ και από την, τελευταία, από την εμπειρία μας των τελευταίων μηνών πρέπει να πω ότι η Ισπανική Προεδρία έχει φροντίσει πάρα πολύ τα θέματα της δικής μας ε, Επιτροπής. Είχαμε πολλές προσκλήσεις, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τις ε, πληρώσουμε όλες, αλλά θεωρώ ότι και τα θέματα πολιτισμού εκπαίδευσης αλλά και τα θέματα αθλητισμού είναι σε πολύ καλά χέρια στα χέρια του Υπουργού. Να σας θυμίσω μόνο ότι κατά τη διάρκεια της ε, θητείας σας ως ε, Προεδρεύοντος του Συμβουλίου ε, αναλύθηκαν αρκετές ε, σημαντικές πρωτοβουλίες. Τώρα κατά πόσο αυτές θα καταλήξουν σε κάποιο μέτρο εφαρμόσιμο θα το δούμε. Μιλούμε για την κοινωνική διάσταση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Μιλούμε για την υποστήριξη της ε, διαβιομάθησης, για, τις, ιδιαίτερες, για τα προσόντα για τις θέσεις εργασίας. Επίσης συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και της ε, οικονομίας, του κλάδου, της βιομηχανίας. Ε, πολύ σημαντικά θέματα λοιπόν που έχουν να κάνουν και με την στρατηγική για το 2020. Ελπίζω αυτό που ανέλαβε η Προεδρία του Συμβουλίου να μειώσουμε δηλαδή την, ε, τα παιδιά που φεύγουν από το σχολείο από 15% σε 10% ε, και να υπάρχει μεγαλύτερη εγγραφή σε υψηλά σε ε, ιδρύματα τρίτης βαθμίδας εκπαίδευσης, να αυξηθεί αυτό στο 40%. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ο κύριος Υπουργό έχει το λόγο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, έρχομαι για δεύτερη φορά εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας και Νεολαίας για να κάνω τον απολογισμό της Ισπανικής Προεδρίας σε θέματα παιδείας και κατάρτισης. Στη διάρκεια αυτών των έξι μηνών συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα κράτη-μέλη, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες, με διάλογο και συνένεση, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για την δέσμευσή τους και την ε, αδιαμφισβήτητη διάθεσή τους να εργαστούν για τη βελτίωση της ε, παιδείας και της επιμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδη ε, της ε, Ευρωπαϊκής Προεδρίας είναι ε, χάρη σε όλους και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είναι συλλογικές επιτυχίες. Θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας σε θέματα παιδείας από την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ μέχρι το ψήφισμα στην Ολομέλεια στις 16 Ιουνίου του 2010 για τη στρατηγική του 2020. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ζούμε στιγμές ε, δύσκολες ε, ως συνέπεια της σοβαρής οικονομικής κρίσης και η έξοδος από την κρίση είναι η μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Από εδώ προκύπτουν και δύο μεγάλοι στόχοι της Ισπανικής Προεδρίας. Πρώτον, δηλαδή, να ε, ξεκινήσει η ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και των θεσμών που δημιουργούνται από τη Συνθήκη και δεύτερον, να ενισχύσουμε τον οικονομικό συντονισμό στα πλαίσια της Ένωσης προκειμένου να καταπολεμήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο την κρίση και να δώσουμε όθηση για την ανάκαμψη. Θα πρέπει να ξεκινήσει οριστικά ένα νέο στάδιο στην ε, νομισματική και οικονομική ε, ένωση που συνεισφέρει αποφασιστικά στη σταθερότητα και στην πρόληψη μελλοντικών κρίσεων. Η Ισπανική Προεδρία με πολύ συγκεκριμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση δεσμεύτηκε προκειμένου να προχωρήσει σε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο θα είναι πιο ε, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο. Ένα μοντέλο στο οποίο η παιδεία και η κατάρτιση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινωτικών πολιτικών. Όταν προ... Το ήρθα στην Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου, σας ανακοίνωσα ότι η Ισπανική Προεδρία θα έβαζε τις αξίες της παιδείας πάνω από όλες ε, τις πιο ε, θεσμικές συζητήσεις. Σκεφτόμαστε με την Ευρώπη, αλλά κυρίως ε, σκεφτόμαστε τους πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες και για αυτούς και για αυτές εργαστήκαμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε μία έθωση στην παιδεία και να την έχουμε στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών. Η παιδεία και η επιμόρφωση είναι ο βασικός πυλώνας της προσωπικής και επαγγελματική ανάπτυξης των πολιτών και γι' αυτό είναι απαραίτητος για την κοινωνική συνοχή και για την ευημερία. Η παιδεία είναι απαραίτητη για να μπορεί κάποιο να είναι ενεργό πολίτη. Η παιδεία είναι το στοιχείο το οποίο εγγυάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ισότητα των ευκαιριών. Η παιδεία είναι το καλύτερο όπλο στη μάχη κατά τη ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι πράγματι η καλύτερη κοινωνική πολιτική. Τον Ιανουάριο Σα παρουσίασα μια σειρά από στόχου της Ισπανική Προεδρία στον τομέα τη παιδείας και τη επιμόρφωση που συγκεκριμενοποιούνται σε τέσσερις βασικέ προτεραιότητε. Να βρίσκεται η παιδεία στο επίκεντρο τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση τη παιδείας και τη κατάρτιση, Να προάγουμε τις βασικές δεξιότητες ε, για την υποστήριξη της κατάρτισης και την υποστήριξη νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις απασχόλησης. Να δώσουμε την όθηση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Γνώσης ως σύγκληση των δύο μεγάλων χώρων στην Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, τον Ευρωπαϊκό Χώρο της ανώτατης εκπαίδευση και τον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας, εξυγχρονίζοντα και διεθνοποιώντας τα πανεπιστήμια μας. Τώρα που τελειώνει η Ισπανική Προεδρία, ήγει και η ώρα να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε τον απολογισμό μας. Και γι' αυτό ακριβώς βρίσκομαι εδώ σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσία των εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών το κοινοβούλιο είναι ο χώρος ε, στον οποίο ε, εκφράζεται με ε, πολύ σοβαρό τρόπο η εμπιστοσύνη στο διάλογο. Εδώ μιλάμε και ακούμε. Έχουμε αντιπαράθεση ιδεών που φέρνει αποτελέσματα και έχουμε ωφέλη από τη συζήτηση. Μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία από τη διάσταση απόψεων ο απολογισμό ενώπιον των πολιτών δεν είναι μόνο υποχρέωσή μα, αλλά είναι και απαραίτητη συνθήκη για να υπάρχει δημοκρατία. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ σήμερα και είμαι πεπισμένο ότι μιλάω στα 500 εκατομμύρια πολίτε ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θα σα αναφέρω τι πρόοδοι έχουν επιτευχθεί για του στόχου που σα ανέφερα ε, προηγουμένως. Πρώτον, το να βρίσκεται η παιδεία στο επίκεντρο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Το να βρίσκεται η παιδεία στην καρδιά αυτής της ε, στρατηγικής ήταν ο μεγάλος στόχος της ε, Ισπανικής Προεδρίας. Η παιδεία δεν ήταν τμήμα των μεγάλων ε, κοινοτικών πολιτικών. Υπήρχε μεγάλη συνένεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν η Ευρώπη θέλει να οικοδομήσει ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, το οποίο θα είναι πιο βιώσιμο, πρέπει να προωθήσει την κοινωνία της γνώσης και να δώσει ευρωπαϊκή όθεση στην παιδεία, στην κατάρτιση, στον πολιτισμό, την καινοτομία και την ε, μεταφορά όλων αυτών στην κοινωνία. Από την αρχή της Προεδρίας μας ε, προωθήσαμε αυτή τη συζήτηση για το ρόλο που θα πρέπει να έχει παιδεία και κατάρτιση στη νέα στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Συνεργαστήκαμε μονίμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, προετοιμασία αυτής της στρατηγικής και η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μετά από τη συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας το Φεβρουάριο έδινε έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθεί η παιδεία και η κατάρτιση στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να αποτελεί συνολικό στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής με στόχο να βγούμε από την ε, κρίση με βιώσιμο και διαρκή τρόπο ως ε, προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας ε, παρουσιάσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη θέση μας, ε, στην οποία επισημαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της παιδείας και της κατάρτισης στη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της το Μάρτιο για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 καθόρισε μία σειρά από βασικές πρωτοβουλίες πολλές από αυτές ε, άμεσα συνδεδεμένες με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ένωση για την καινοτομία, νεολαία για την μετακίνηση, μία ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη και μία ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και τις θέσεις απασχόλησης. Και από κοινού με αυτές τις θέσεις ε, το Ευρωπαϊκό ε, Αρινό Συμβούλιο συζήτησε ένα πρώτο κείμενο για τη νέα στρατηγική και καταλήξαμε σε μία συμφωνία για τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να την αποτελούν, περιλαμβανομένων και των πέντε βασικών στόχων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και αυτός ο οποίος σχετίζεται με τη βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και κυρίως με το στόχο να μειώσουμε την εγκατάλειψη του σχολείου και να αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που ολοκληρώνει τις ανώτατες ε, σπουδές ή κάποιο αντίστοιχο επίπεδο ισοδύναμο. Στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Παιδεία του Απριλίου, ε, οι Υπουργοί επανέλαβαν αυτή τη σημασία του ρόλου της παιδεία και τη στρατηγική και το πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθούν αυτά τα ποσοστά ε, μέχρι το 2020. Στο Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργών Παιδεία του Μαΐου η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεισφορά ε, στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην οποία είχαμε δώσει τον τελικό ρόλο να καταλήξει στις συμφωνίες για τη στρατηγική του 2020. Ε, υπ' αυτή την έννοια, με σκοπό να βελτιώσουμε την παιδεία της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία, ε, τέθηκε το γεγονός ότι πρέπει να μειώσουμε το ποσοστό της εγκατάλειψης του σχολείου στο 10% κατά μέγιστο και να αυξήσουμε κατά 40% το ποσοστό του πληθυσμού που ε, λαμβάνει ανώτατη εκπαίδευση ή κάποια αδύναμη εκπαίδευση τότε οι 26 από τα 27 κράτη-μέλη υποστήριξαν αυτά τα αριθμητικά ποσοστά, παρά το γεγονός ότι δυστυχώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπόρεσε να υποστηρίξει, διότι ε, ε, βρισκόταν σε φάση σχηματισμού νέας κυβέρνησης, αλλά η συμφωνία στην οποία ε, καταλήξαμε το Συμβούλιο, 26 εκ των 27 κρατών, υλο, ε, από εκεί και πέρα μεταφράστηκε σε συμπεράσματα της Προεδρίας και όχι του Συμβουλίου, ε, διότι χρειαζόμαστε ομοφωνία. Εν τέλει, και αυτό είναι καλό νέο για όλους, ε, από την Προεδρία μεταβιβάστηκαν αυτά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση που είχαμε στις 17 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε πέντε ποσοτικούς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε θέματα απασχόλησης, παιδείας, καινοτομίας, Αλλαγή του κλίμακος και κοινωνική ένταξη. Μου φαίνεται ότι είναι καλά τα νέα αν η παιδεία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ αυτών των στόχων και θεωρώ ότι είναι καλό το αποτέλεσμα δεδομένου ότι αυτή η παιδεία αφορά ε, εγκάρσε και τους υπόλοιπους στόχους. Σε θέματα παιδείας καθορίστηκαν οι δύο ποσοτικοί στόχοι που σας ανέφερα πριν και μάλιστα με τα ποσοστά που είχαμε προτείνει εμείς. Επομένως, για πρώτη φορά η επαιδεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ κυρίες και κύριοι ότι θα πρέπει να συγχαρούμε αλλήλους ε, για τον στόχο αυτό, διότι εδώ και χρόνια εργάζεστε και εργαζόσαστε για αυτό το θέμα και για πρώτη φορά υπάρχει βούληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί ένα νέος δεσμός μεταξύ οικονομίας και παιδείας. Ένας δεσμός ο οποίος ενισχύει την ιδέα της κοινωνικής Ευρώπης, διότι θέτει την ε, παιδεία στο επίκεντρο της οικονομίας. Για πρώτη φορά η Ευρώπη γράφεται με το ε της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι εργαστήκαμε πολύ καλά και για πολλά χρόνια και εμείς ήμασταν απλώς αυτοί οι οποίοι αναλάβαμε το ρόλο και θέλαμε να καταδείξουμε τα αποτελέσματα των εργασιών σας. Δεύτερον, θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της παιδείας και της κατάρτισης. Κυρίες και κύριοι, όπως σας έλεγα πριν, η παιδεία είναι το καλύτερο ε, στοιχείο για την κοινωνική ένταξη. Οι ίσες ευκαιρίες σημαίνουν ότι υπάρχει και ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία. Σήμερα είναι περισσότερο απαραίτητο από ό,τι ποτέ, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει θέσει σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού πληθυσμού πολλούς πολίτες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, από την αρχή της Προεδρίας, θέσαμε την κοινωνική διάσταση της παιδείας ε, στον κεντρικό άξονα των προτάσεων, των συζητήσεων και των καθηκόντων μας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, συγγνώμη, στο Συμβουλίο Παιδείας του Φεβρουαρίου έγινε μία άτυπη συζήτηση για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική διάσταση της παιδείας και της κατάρτισης και τα κράτη-μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους για να υπάρχουν ε, πολιτικές ε, παιδείας που θα περιλαμβάνουν περισσότερους και θα είναι πιο ισότιμες και μεγαλύτερες ποιότητες. Στο Συμβούλιο Παιδείας του Μαΐου, μετά από μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στην ανάλυση των τρόπων με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε του κινδύνους της ανεργίας και του αποκλεισμού, οι Υπουργοί υιοθέτησαν ένα έγγραφο συμπερασμάτων για την κοινωνική διάσταση της παιδείας και της κατάρτισης. Εκεί καλούνται τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα για να διευρυνθεί η πρόσβαση σε παιδεία υψηλής ποιότητας ε, τονίζοντας κυρίως ένα ε, σύστημα ε, παιδικής παιδείας ποιότητας. Γι' αυτό προτείνεται να υπάρχουν οι βασικές δεξιότητες στο δημοτικό σχολείο, κυρίως η ανάγνωση και τα μαθηματικά. Βασικές αξίες για να μπορέσει να δοθεί όθηση και να αποκτηθούν οι βασικές δεξιότητες για τους ενήλικες. Η ολοκλήρωση των, και ενσωμάτωση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα γενικά συστήματα μέσω ευέλικτων οδών, καθώς επίσης και να διευρύνουμε την, την πρόσβαση και την ανώτατη διδασκαλία όλων των φοιτητών με οικονομική στήριξη και ευέλικτες δυνατότητες για να μπορούν να εγγυηθεί σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ενηλίκων, ότι θα έχουν πρόσβαση σε βασικές δεξιότητες. Θεωρώ ότι υπάρχει συνένεση και είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα θέλουν να διασφαρίσουν κοινωνική ισότητα και ακαδημαϊκή αριστεία διότι η ισότητα και η αριστεία δεν αποκλείουν κανέναν. Είναι αρχές οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και περιλαμβάνουν τους πάντες. Τρίτον, θέλουμε να αναπτύξουμε τις ε, ε, αρμοδιότητες για υποστήριξη τη μόνιμη κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση, νέες δεξιότητες για νέες θέσεις απασχόλησης. Κυρίες και κύριοι, όταν ήρθε εδώ τον Ιανουάριο, σας ανέφερα ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα στενός δεσμός μεταξύ παιδεία και απασχόληση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν θέσει εργασία οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μία ε, αένεη διαδικασία. Πολλοί μπορεί να αλλάξουν πολλές θέσεις εργασίας στη διάρκεια της ζωής τους και πολλές ε, γνώσεις που θα αποκτήσουν θα είναι οι δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές και στην ε, ολοένα αυξανόμενη ευελιξία των αγορών εργασίας. Μεταξύ των εργασιών λοιπόν της Επιτροπής Παιδείας ε, στο ε, Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας το Μάιο υιοθετήσαμε κάποια συμπεράσματα για τις ε, ε, δεξιότητες προς υποστήριξη της διαβίου κατάρτισης. Ο τίτλος ήταν «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις απασχόλησης» και σχετίζεται στενά με τους στόχους για την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Αυτή η στρατηγική καθορίζει ότι η Ευρώπη ε, στο μέλλον και με τις εργασιακές και επαγγελματικέ της προοπτικές ε, θέλει να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπινους πόρους και να ε, επικαιροποιήσει τις απαραίτητες αρμοδιότητες. Η δέσμευση που υιοθετήσαμε ως κράτη-μέλη συγκεκριμενοποιείται με απόκτηση, επικαιροποίηση και ανάπτυξη των βασικών αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της παιδείας και της κατάρτισης. Να ετοιμάσουμε τους ε, διδάσκοντες, ε, τους όσους κάνουν κατάρτιση και τις διευθυντικές ομάδες για αυτή τη μεγάλη αλλαγή και να προσεγγίσουμε τον εκπαιδευτικό κόσμο και τον κόσμο της κατάρτισης με τον γενικότερο κόσμο, κυρίως τον κόσμο της εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο και να αξιολογήσουμε τις δεξιότητες που αποκτούμε ε, με άτυπο ή με επίσημο τρόπο. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύονται να υποστηρίξουν την επαγγελματική ανάπτυξη, την αρχική και τη μόνιμη όλων όσων συμμετέχουν στον εκπαιδευτικό κόσμο και στον κόσμο τη κατάρτιση, καθώ επίση και να ενδυναμώσουν την εργασία σε συνεργασία με του κοινωνικού εταίρου και με τι ε, δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση για να μπορέσουν να προσεγγίσουν την παιδεία και την κατάρτιση με τις επιχειρήσεις και τους ε, εργοδότες. Τέταρτος στόχος, διεθνοποίηση και εξυγχρονισμός της ανώτατης ε, παιδείας. Η ανώτατη παιδεία θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, βελτίωση τη κοινωνική ευημερία και το οικονομικό μα μέλλον. Στη αρχή τη Ισπανική Προεδρία αποφασίσαμε να εμβαθύνουμε στον ευρωπαϊκό χώρο τη ανώτατη εκπαίδευση και να προχωρήσουμε την ατζέντα εξυγχρονισμού των πανεπιστημίων που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Συμβούλιο Υπουργών του Μαΐου υιοθετήθηκε ένα συμπέρασμα το οποίο θεωρείται θεμελιώδε και θέλουμε να καθορίσουμε σχέσεις και με τρίτες χώρες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ανταλλαγές ταλέντου και να κυκλοφορούν οι εμπειρίες. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια αυθεντική ε, διεθνή κουλτούρα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυξάνοντας τις δραστηριότητές τους και την παγκόσμια διάστασή τους. Θέλουμε να προάγουμε τη διεθνή διάσταση και την κοινωνική ευθύνη των πανεπιστημίων μέσω τη συνεργασία και μέσω των ε, διαφόρων ανετάτων ιδρυμάτων των διαφόρων χωρών, εγγυόμενη την ε, ισότιμη πρόσβαση στου πολίτε, ε, στα πανεπιστήμια και στην κινητικότητα. Επίση, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική προ αυτή την κατεύθυνση που θα συντονίζει τι διάφορε πρωτοβουλίε που ήδη είναι ενισχύ και θα προάγει την διεθνή προβολή τη ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτά τα συμπεράσματα καλούμε επίσης τις χώρες μέλη να δώσουν κίνητρα για την επιστροφή της γνώσης στην κοινωνία, για να εμβαθύνουμε στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης παιδείας και να καθορίσουμε ένα νέο πλαίσιο για το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού χώρου της γνώσης. Τέλος, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ισπανία είχε την ε, συμπροεδρία των ε, συνεδριάσεων της Υπουργικής Διάσκεψης της Βουδαπέστης Βιέννης και της ε, συνεδριάσεις της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Πολώνια. Ε, και τα αποτελέσματα θα πρέπει να υπερτονιστούν εδώ. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Υπουργική Διάσκεψη Βουδαπέστης Βιέννης. Ναι. Επιπλέον, οι συνεδριάσεις της Ομάδας Παρακολούθησης στην Πολώνια και στην Υπουργική Διάσκεψη ε, έγιναν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να τονίσουμε το μέτρο για την διεθνή κινητικότητα των φοιτητών, ε, με το κριτήριο που καθορίζεται στη δήλωση της ε, Λοβαϊνά που λέει ότι το 2020 τουλάχιστον το 20% των πτυχιούχων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν θητεύσει ή να κάνουν πρακτική εκπαίδευση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, καθώς επίσης και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Προαγωγής και Ενημέρωσης ε, του Ευρωπαϊκού Χώρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ναι. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάποια επιπλέον σημεία τα οποία έχουν ε, ε, σχέση με την έναρξη της συζήτησης για τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πριν ε, ολοκληρώσω, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι πέραν των προηγούμενων συμφωνιών ξεκινήσαμε και προωθήσαμε κάποια άλλα στοιχεία για τον τομέα της παιδείας. Καταρχά, θα ήθελα να σα επισημάνω την έναρξη τη συζήτηση για το συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα γενεά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ε, για να ε, τα συνδυάσουμε με την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Η άτυπη Σύνοδο Υπουργών Παιδεία του Απριλίου συζήτησε τη νέα γενεά ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπό το φως της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 και παρά το γεγονό ότι αντιπροσωπείε ε, τόνισαν ότι επετέφθηκαν Υπάρχουν ε, πολύ καλά πράγματα ε, μέχρι τώρα με τα διάφορα υποπρογράμματα του προγράμματος ε, διαβίου μάθηση. Το αρχικό συμπέρασμα ήταν ότι ε, δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποκαταστήσουμε τα προγράμματα τα οποία αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, αλλά απλώς να τα ενδυνασμώσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινού τόπους για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η νέα στρατηγική. Καταρχά επιμείναμε στο γεγονό ότι η πρωτοβουλία νεολαία ε, και μετακίνηση θα πρέπει να χρησιμεύσει για να μπορέσουμε να αυξήσουμε του δεσμού μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων και τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 και με τι πολιτικέ ε, νεολαία και απασχόληση και ταυτόχρονα επισημάναμε πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν σε αυτέ τι δράσει, οι νέοι φοιτητέ και όλοι όσοι ενδιαφέρονται, ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οικονομικοί και κοινωνικοί φορεί και εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών δεν θέλουμε απλώς ε, να συνεργαστούμε για αυτούς, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Ολοκληρώνω κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εξάμεινο σκληρής δουλειάς, το οποίο θεωρώ ότι μας βοήθησε για να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει σε θέματα παιδείας. Πρόκειται για ένα καθήκον το οποίο φυσικά δεν ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Η Προεδρία είναι πάντα περαστική. Οι επόμενες Προεδρίες, κυρίως η Βελγική και η Ουγγρική, ως ε, μέλη του τρίου, θα πρέπει να εμβαθύνουν στην ανάπτυξη αυτών των μεγάλων ε, στόχων που καθορίστηκαν στη στρατηγική του 2020. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους ε, για τα όσα έκαναν και για το γεγονός ότι διευκόλυναν το έργο της Προεδρίας και θα ήθελα να επαναλάβω, για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω στην Επίτροπο κυρία Βασιλείου και στα κράτη-μέλη και όλους εσά για τη βοήθειά σα και την αφοσίωσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ακούγοντά σα. νόμιζα ότι σύντομα θα τελειώσει ο παράδεισος. Όλες αυτές οι ωραίες λέξεις, οι ωραίες κουβέντες που μας είπε ο υπουργό, αν οδηγούσαν κάποτε σε ένα σχέδιο εφαρμόσιμο θα ήταν πολύ ωραία. Ξέρω ότι εσείς είσαστε μόνο ένας από τους 27 και ο κάθε ένας από τους 27 πρέπει να παραδεχτεί τα λάθη του. Αλλά αν μιλάμε για μια προεδρία, τότε θεωρώ ότι τον επόμενο χρόνο ακόμα την ίδια έμφαση θα δίδει σε αυτή τη δουλειά, στην εργασία. Και ελπίζω να έχουμε τελικά τα προγράμματα τα πολιτιστικά, τα εκπαιδευτικά, τα προγράμματα για τον αθλητισμό που χρειαζόμαστε. Ελπίζω κύριε Υπουργέ να έχουμε διαθέσιμα αυτά τα προγράμματα κάποια στιγμή. Εγώ σας εμπιστεύομαι πάντως. Η κυρία Χάνιβαλ έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας εξηγήσατε με τέτοια λεπτομέρεια και τόσο σαφώς τα θέματα που απασχολούν την Ισπανική εδρία Και είναι πολύ θετικό ότι δίνεται τέτοια προτεραιότητα στην παιδεία και εμείς στην Επιτροπή μας ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για αυτήν. Πολλά από αυτά που συστήνεται είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επαγγελματική επιμόρφωση, πρόσβαση. Εξαιρετικά επαναλαμβάνω είναι όλα αυτά, αλλά θέλω να θέσω και ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κυβερνήσεις χρειάζεται να κάνουν περικοπές σε όλες τους τις δαπάνες. Πώς βλέπετε την προτεραιότητά σας για την παιδεία να εφαρμόζεται με τέτοιες συνθήκες. Δούμε. Μπαρούνια Μπάνια Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ στην αίθουσα, στην Επιτροπή μας. Όταν ήρθατε στην αρχή της Ισπανικής Προεδρίας και για να μας παρουσιάσετε τους στόχους σας, ε, το είχα εκτιμήσει ιδιαίτερως και θα ήθελα να πω ότι ενθουσιάστηκα από τη δέσμευσή σας και από το γεγονός ότι, όπως είπατε εσείς, η παιδεία βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της Προεδρίας. Ναι, ναι, ναι. Με χαροποιεί επίσης το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος ε, συντονισμός μεταξύ των προτάσεων που μας ε, αναφέρατε με τους ε, στόχους ε, της Επιτροπής μας. Παρατηρώ μια σύμπνοια. Διάβασα εδώ κάποια σημειώματα για το Συμβούλιο του Μαΐου και πραγματικά είναι απόλυτη η σύμπνοια. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι για μένα ένας από αυτούς τους στόχους που βρίσκεται στις αποφάσεις είναι ίσως ε, κατ' εμέ ο πιο σημαντικός. Και είναι αυτός των νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις απασχόλησης. Θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα κρατημέλη, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και αυτό είναι η ανεργία των νέων. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας και νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με καλύτερη επιμόρφωση και καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον. Κατανοώ αυτά που μόλις είπε η κυρία Χάνιμπολ και συμμερίζομαι και εγώ τις απόψεις της, διότι βιώνουμε χαλεπούς καιρούς, επομένως θα χρειαστούμε να χρησιμοποιήσουμε και πόρους, αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι ένας από τους στόχους που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε. Και επίσης ε, ελπίζω ε, η δέσμευση της Προεδρίας αυτής για την παιδεία να συνεχιστεί και για τις επόμενες Προεδρίες, και τη Βελγική και την Ουγγρική, και να μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις μεγάλες προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ. Σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ζητώ συγγνώμη, ήρθα λίγο καθυστερημένο, δεν μπόρεσα να ακούσω την αρχή τη παρουσίασή σα. Ευχαριστώ για τι πληροφορίε που μα δώσατε. Θα ήθελα να σα κάνω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει. Στο θέμα της διαδικασίας της Μπολόνια αναφερθήκατε στην κινητικότητα των ε, μαθητών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμένα μου φαίνεται θεμελιώδες, αλλά η διαδικασία του Μπολόνια ε, συζητά και το θέμα της κινητικότητα των καθηγητών. Θα ήθελα να ξέρω αν έγινε κάποια πρόοδο επί του θέματο αυτού, σε θέματα κινητικότητα καθηγητών, διότι ορισμένε φορέ είναι πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν έδρε ε, και δεν είναι τόσο εύκολη μετακίνηση, αλλά καλό θα ήταν να μπορούν και οι καθηγητέ να διεξάγουν τι δραστηριότητέ του σε άλλα πανεπιστήμια. Και υπάρχει και ένα ακόμα σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και εμά εδώ στην Επιτροπή μα ενδιαφέρει πολύ. Ο πρόεδρο Μπαρόσο αναφέρεται στην νεολαία και στην κινητικότητα αλλά εμάς μας ανησυχεί και η διαβίου μάθηση. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί μόνο η νεολαία, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντική, θα πρέπει να σκεφτούμε και τους ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας για να μπορέσουν να συνεχίσουν την επιμόρφωση στη διάρκεια όλης της της ζωής. Αυτές τις ερωτήσεις λοιπόν ήθελα να σας κάνω και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ο κύριος Μπερλουγκουέρ. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ε, πειθό που επιδείξατε στα θέματα της διαβίου μάθησης, στην κοινωνία της γνώσης και τους στόχους ε, που ε, είναι εγκάρσιοι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση με βάση και όλα όσα ακούσαμε με την, πρόεδρο μετά, ε, την πρόεδρο μετά τις παρεμβάσεις σας. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εσείς είστε πεπισμένος για αυτά που μας είπατε. Αλλά εμείς ακούμε πάρα πολλά λόγια για την ε, προτεραιότητα της παιδείας και στην πράξη βλέπουμε πάρα πολύ λίγα. Υπερτονίζουμε τα θέματα της παιδείας και όταν φτάνουμε σε θέματα προπολογισμού την έχουμε Στη τελευταία σειρά των επενδύσεων. Με εξέπληξε θετικά το γεγονός ότι η Γερμανία έχει ένα, μια μεγάλη παρέμβαση εξυγίασης, 80 δις ευρώ και το μόνο στοιχείο το οποίο αύξησε στις δαπάνες ήταν το θέμα της παιδείας και της έρευνας. Που σημαίνει ότι όταν θέλουμε να αναζητήσουμε κονδύλια μπορούμε να τα βρούμε. Γιατί λοιπόν δεν καταφέρνουμε να τα υλοποιήσουμε στην πράξη αυτά τα θέματα των προτεραιοτήτων. Γιατί δεν συγκεκριμενοποιείται η παιδεία. Θα ήθελα να σας προτείνω κάτι. Μια ιδέα που μπορεί να είναι πολύ ε, λίγη, μπορεί να είναι λαθασμένη. Θεωρώ ότι δεν έχουμε αναπτύξει επαρκώς ε, τη βαθιά αλλαγή της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μεγάλης αλλαγής που προκύπτει από την τεχνολογία της γνώσης αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε μόνο θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας εξειδικευμένες, χρειαζόμαστε καινοτομία, δημιουργικότητα στα σχολεία για να μεταλαμβαδευτεί αυτό σε δημιουργικότητα στην κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε αυτά στα σχολεία μας. Ένα δεύτερο σημείο, πολύ γρήγορα, αναφερθήκατε στη διαδικασία της Μπολόνια. Ε, πολύ πιστικά επιχειρήματα, τα προσυπογράφω κι εγώ, αλλά γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προσκόμματα στη διαδικασία της ε, Μπολόνια. Πάρα πολλά προσκόμματα. Και πολύ συχνά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ε, απλώς ε, συζητάται στις υπουργικές διασκέψεις κάθε δύο χρόνια και στην πανεπιστημιακή βάση δεν συζητάται επαρκώς. Εμείς πρέπει να επενδύσουμε στα πανεπιστήμια και δεν πρέπει να παρνηθούμε αυτό το στόχο. Θα πρέπει να δοθεί ιδέουσα ενέργεια στα πανεπιστήμια και θα ήθελα να ζητήσω και την άποψη άποψή σας επ' αυτού. Τα πανεπιστήμια πρέπει να εκδίδουν ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών, όχι μόνο εθνικού τίτλου σπουδών και πρέπει να το αναλάβουν το πρόβλημα αυτό. Αν υπάρχουν δυσκολίε, να του βοηθήσουμε να τι επιλύσουν, αλλά να μην οπισθοχωρήσουμε σε καμία περίπτωση. Και αυτό θα ήθελα να σα ζητήσω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τελευταίο ο κύριο Παπα-Νικολάου. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πράγματι η Ισπανική Προεδρία ε, και εγώ πιστεύω έκανε σοβαρή προσπάθεια και σας ευχαριστούμε για όλη αυτή την πορεία. Ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Το πρώτο, σε συνέχεια των όσων υπόθηκαν και από τους συναδέλφους. Αναφερόμαστε στην ανάγκη να ενισχύσουμε τους νέους ανθρώπους και να έχουν νέες ευκαιρίες και να έχουμε σύνδεση της εκπαίδευσης, ειδικά της ανώτατης εκπαίδευσης, με την αγορά εργασίας. Έχουμε ε, το τρίγωνο της γνώσης, όπως το αναφέρουμε και στρατηγική 2020, έρευνα, καινοτομία, ε, εκπαίδευση και μια διαπίστωση που κάνουμε είναι ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, για παράδειγμα, ε, στον τομέα της πληροφορικής θα χρειαστούν περίπου, μας είπε η κυρία Κρός, η Επίτροπος σε μια άλλη συνάντησή μας, περίπου 700.000 θέσεις, νέες, εργασ... θέσεις εργασίας. 700.000. Αυτό το γνωρίζουμε. Στον τομέα της παιδείας προσαρμόζουμε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα ώστε να δώσουμε στους νέους περισσότερες ευκαιρίες μέσα από αυτές τις επιστήμες. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός μας, χρειάζεται ένα συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Αναφερόμαστε συνεχώ σε αυτή την περιβόητη, επιτρέψτε μου, ανοιχτή μέθοδο συνεργασία. Ήμουν ο για την έκθεση για την νεολαία από πλευρά του, της Επιτροπής μας και προσπάθησα να καταλάβω πώ ακριβώ λειτουργεί αυτό. Μετά από αρκετά χρόνια που εφαρμόζεται, εγώ διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και ο συντονισμό ε, δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν μαθαίνουμε τι συμβαίνει σε αυτό το συντονισμό, δεν έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα, Πολλές φορές τα κράτη-μέλη υποβαθμίζουν τα ίδια την παρουσία τους σε αυτή την προσπάθεια και τελικά ειδικά στο θέμα της παιδείας που έχουμε επικουρικότητα και ενώ εμείς λέμε εδώ ωραία πράγματα, ενώ τοποθετούμαστε με συγκεκριμένες πολιτικές, αυτά τελικά δεν φτάνουν σε ένα σημείο αφομοίωσης από τα κράτη-μέλη. Σας ερωτώ λοιπόν ως δεύτερο ερώτημα αν εσείς ως Προεδρία διαπιστώσατε αυτά τα προβλήματα και αν νομίζετε ότι άμεσα πρέπει να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών. So, the last is... Ο κύριος Τσβέρ έχει το λόγο. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod minister, predsednik. Kje je Burge? Καταλαβαίνω μεν τη θέση σας, την κατανοώ. Το 2008 κατά τη Σλοβενική Προεδρία χρειάστηκε και εγώ να κάνω κάτι ανάλογο με εσά και κατανοώ τους φραγμούς που αντιμετωπίζετε στις προσπάθειές σας. Οι στόχοι που μας περιγράψατε στην αρχή του έτους κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της Ισπανικής Προεδρίας ήταν πολύ σημαντικοί και είμαι βέβαιος ότι σήμερα που κάνουμε την αξιολόγηση μπορείτε να είστε ικανοποιημένος. όλα αυτά επιτρέψτε μου να θέσω και μερικά ερωτήματα που πιστεύω ότι αντιμετωπίζει προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή παιδεία σήμερα. Μου φαίνεται ότι δεν αρκεί η καλή θέληση. Έχουμε 8, 8 εκατομμύρια α, θέσεις εργασίας για, οι οποίες δεν πληρούνται από καλά μετεκπαιδευμένους ανθρώπους. Το 1 τρίτο των θέσεων μάλιστα θα μπορούσα να πω σε ολόκληρη την Ένωση δεν πληρεί τα προσόντα που απαιτούνται. Λόγω δε της κρίσης δεν είναι ικανοποιημένη η οικονομική κοινότητα με τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής παιδείας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθωθεί αυτό ώστε οι νέοι ερευνητές επιστήμονες από εκτός, εκτός ενώσεως να μπορέσουν να έρθουν και αυτοί να ελκυστούν εδώ. Η γύρανση του πληθυσμού σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι υλικό διαθέτουμε και όχι μόνο τους νέους. Θα μπορούσαν να μπορούσαμε να φανταστούμε και άλλες λύσεις, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολες να εφαρμοστούν, όπως τον καθορισμό με ενό νέου τύπου παιδείας για τη νέα μεταβιομηχανική εποχή όπου να απαιτούνται νέα προσόντα και νέες μέθοδοι και θέματα διδασκαλίας. Στην ανώτερη εκπαίδευση, στην Ένωση δεν τα πάμε άσχημα, αλλά σε επίπεδο της διαδικασίας της Βολονίας έχουμε αποτύχει. Η διαδικασία αυτή είναι ανεπαρκής, ανεπιτυχής και τα κράτη-μέλη δεν επενδύουν αρκετά για να βελτιώσουν την πρόσβαση των μαθητών και φοιτητών στην ναι, αυτή η διαδικασία. Είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσά που διαθέτουμε από ό,τι στις Ηνωμένε και την Ιαπωνία και τώρα που γίνονται και νέες περικοπές ακόμη και στην παιδεία πρέπει να παραδεχτούμε ότι ζούμε σε πολύ περίεργες εποχή, πολύ περίεργη εποχή. Μπορεί πολλοί να μην θέλουν πια καν την παιδεία ενώ είναι τελείως απαραίτητη αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε οι ίδιοι. Βέβαια πρέπει μονίμως να γίνεται εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Συμφωνώ και με τον κύριο Παπα-Νικολάου που είπε ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού ή συνεργασίας δεν αρκεί πια για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Ίσως να, χρειάζεται μια, δύο, να χρειάζονται μια-δυο οδηγίες για αυτό το θέμα. Θα φανεί όμως αυτό. Ούτως ή άλλως ή οπωσδήποτε πιστεύουμε ότι η επόμενη Προεδρία, η Βελγική, θα προσπαθήσει όπως και εσείς να αναζωογονήσει αυτό το θέμα των νέων προσόντων που απαιτούνται για την πρόσβαση στην εργασία, ώστε τα εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη να είναι συγκρίσιμα με των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να μπορούμε και εμείς να έχουμε μια ανάπτυξη ανθρώπινη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ευρύ το φάσμα των ε, ερωτήσεων. Ε, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι μπορείτε απαντήστε. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, αλλάζει η νοοτροπία μας και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την παιδεία. Η κρίση ποτέ δεν είναι καλή, αλλά με την κρίση μάθαμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και εις βάθος η εκπαίδευση διδάσκει, αλλά πρέπει και η εκπαίδευση να μάθει. Και εμείς μάθαμε κάποια πράγματα. Αυτός που δεν έμαθε αυτό το μάθημα θα πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα. Πάρα πάρα πολύ ακριβά, διότι η επένδυση στην παιδεία είναι ακριβή, αλλά το να μην επενδύσουμε στην παιδεία είναι πανάκριβο. Το να επενδύσουμε στην ποδία στοιχίζει, αλλά αν δοκιμάσετε, όπως είπε κάποιος, ε, να επενδύσετε στην άγνοια, θα δείτε πραγματικά πόσο ακριβά στοιχίζει. Κάποιες χώρες αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται αυτό και γνωρίζουν ότι ακριβώς επειδή βρισκόμαστε ε, εντό της οικονομικής κρίσης, που είναι και κοινωνική και πολιτική και κρίση αξιών, Ακριβώς για αυτό το λόγο, περισσότερο από ποτέ, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Και φυσικά δεν αρκεί να είμαστε πεπισμένοι, πρέπει να είμαστε πιστικοί, κάτι το οποίο διαφέρει λίγο και για αυτόν ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ανθρώπους με πολιτικό θάρρος, ε, κοινωνικό θάρρος για να προασπίσουν με καλά επιχειρήματα το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν υπάρχει πραγματικά άλλη διέξοδος ε, για την ε, κρίση από την διέξοδο που προσφέρει η επιστήμη, η έρευνα, η κατάρτιση, η παιδεία, ο πολιτισμός. Αν κάποιος από τους παριστημένους γνωρίζει κάποια άλλη άγουσα, σας παρακαλώ να το πει. Διότι αυτός είναι ο δρόμος. Αυτό το κατανόησαν 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι εγκρίναμε κάποια ε, ψηφίσματα ομόφωνα και 27. Ακούσαμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές, ε, παρά το γεγονός ότι αυτή η ανοιχτή μέθοδος ε, συντονισμού είναι ανεπαρκής, παρά το γεγονός ότι ο καθένας προσπίζεται και τα δικά του συμφέροντα, ε, συνειδητοποίησαμε όλοι ότι η κρίση είναι κοινή και μας αφορά όλους και εγκρίναμε ομόφωνα κάποια θέματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ επίσης ότι πέραν του της αναζήτησης χρηματοδότησης, της αναζήτησης πόρων και της αναζήτησης επενδύσεων ε, στην παιδεία, ε, έχει σημασία να γίνουν και κάποιες συζητήσεις. Συζητήσεις οι οποίες θα είναι συνεκτικές και θα ενδιαφέρουν το θέμα ναι, εντάξει, δεν έχουμε πόρους, αλλά ορισμένες φορές δεν συζητάμε κιόλα. Μας λείπει ο διάλογος. Δεν έχουμε χρηματοδότηση, ορισμένες φορές δεν έχουμε και επιχειρήματα. Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω εδώ είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πιστέψαμε ότι δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο αν κάνουμε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε να ε, παρουσιάσουμε... Ε, χειροπιαστά επιχειρήματα και να βρεθούμε ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών και να μην τους πούμε ότι η παιδεία δεν είναι μια παράπλευρη ιστορία, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μας ενδιαφέρουν οι δημόσιες δαπάνες, σαφώς μας ενδιαφέρει και η κρίση, αλλά αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνώσεων των 27 χωρών μελών αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διαπιστώσουν και το έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία θα πρέπει να εκφραστούν στον προπολογισμό, ελπίζω όταν θα εγκρίνουμε του επόμενου προπολογισμού, θα υλοποιηθούν και θα αποδείξουν αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Πράγματι, Χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας, διότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ε, μας ε, παρακινεί καταπηγόντως να βελτιώσουμε τις ε, κατάλληλες δεξιότητες για τις τέσσερις εργασίες για να βρεθεί η Ευρώπη στο νέο δρόμο της ανάκαμψης. Αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και τις απαιτήσει της κοινωνίας, όχι μόνο τις απαιτήσει της αγοράς, αλλά και όλη την κοινωνία. Ναι. Και χρειαζόμαστε μια οικονομία που, θα έχει, που είναι χαμηλή σε κατανάλωση άνθρακα. Θα πρέπει να διαδοθούν τεχνολογίες πληροφορικής, τεχνολογίες επικοινωνίας, νανοτεχνολογίας. Όλα αυτά μας προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για να δημιουργήσουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η απώλεια πολλών θέσεων εργασίας που σχετίζονται με δραστηριότητες που δεν είναι τόσο παραγωγικές, ε, όπως για παράδειγμα ο κατασκευαστικός τομέας, οι κοινωνικέ υπηρεσίες, ο τουρισμός, κατέδειξαν πόσο λίγες δυνατότητες προόδου υπάρχουν. Ο μας λέει ότι το 2020 το 85% των θέσεων εργασίας θα είναι θέσεις με προσόντα. Επομένως, εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες δεξιότητες, δεν θα υπάρχει ούτε δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης, ούτε ε, απασχολησιμότητα. Και φυσικά, το θέμα είναι επίγον και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι είμαστε πεπισμένοι ότι η μόνη μας δυνατότητα είναι η ε, επαγγελματική εξειδίκευση ε, όσον αφορά την ανεργία των ε, νέων είναι ανησυχητικά τα αποτελέσματα διότι υπάρχουν ε, κάποιοι νέοι που δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση από την παιδική ηλικία διότι η παιδική ηλικία είναι ε, η κατάλληλη στιγμή για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις κατάλληλες δεξιότητες στο σχολείο δεξιότητες, όχι μόνο γνώσεις δεξιότητες ε, για τη βιωσιμότητα της αγοράς εργασίας και κυρίως ε, να γνωρίζουμε βασικά πράγματα, ε, ανάγνωση, γραφή, αριθμητική. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση ε, με τον ίδιο τρόπο που επισημάνατε κι εσείς. Ο κύριος Φίσας μας μίλησε για την κινητικότητα και σαφώς θα πρέπει να μιλάμε και για την κινητικότητα των καθηγητών. Ε, το Μάιο εγκρίθηκε ε, ένα σχέδιο συμπερασμάτων που καθόρισε ως μία από τις προτεραιότητες ε, την κινητικότητα και συμφωνώ, έχετε δίκιο. Αλλά τα συμπεράσματα για τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων που υιοθήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 Μαΐου ζητούν από τα κράτη-μέλη να ε, θεμελιώσουν και να υποστηρίξουν αυτή την κινητικότητα, προσφέροντας τις κατάλληλες δεξιότητες να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στη διαδικασία. Διότι υπάρχει πολλή κινητικότητα, ορισμένες φορές όμως είναι ατομική κινητικότητα που σχετίζεται με τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά δεν είναι επιστημονικές ή πανεπιστημιακές έρευνες και θα πρέπει να τα προωθήσουμε όλα αυτά τα θέματα των πανεπιστημίων και θέλουμε να έχουμε και διεθνείς ε, προοπτικές και ένας από τους άξονες θα πρέπει να είναι και η κινητικότητα των διδασκόντων. Όντως, όταν μιλάμε σε συνεδριάσεις, ε, μιλάμε για κάποιες αρχές, ε, μας τις επεσήμανε και η πρόεδρος, είναι πολύ ωραίες ιδέες όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα υλοποιήσουμε στην πράξη. Προεδρία έχει να σας πει ότι για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού με τη νέα στρατηγική θα πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τα ποια συμπεράσματα ε, υιοθετήσαμε για το γεγονός ότι εγκαταλείπουν τα παιδιά νωρίς στο σχολείο και ένα 10% θα πρέπει να είναι το μέγιστο όριο. Αλλά το θέμα είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την απόφαση. Πώς θα την παρακολουθήσουμε την απόφαση που υιοθετήθηκε. Κάθε φορά που υιοθετείται κάτι στην Ευρώπη, ε, κάποια συμπεράσματα, περνάει ο καιρό και διαπιστώνουμε ότι μετά δεν τα τηρήσαμε. Και νομίζω ότι ένα από τα πιο βασικά σημεία αυτή τη στιγμή είναι ε, η διακυβέρνηση της ε, εξέλιξης και της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχουμε ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τους στόχους της στρατηγικής για το 2020. Η διαδικασία της Μπολόνια είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Επιτρέψτε μου ε, βρισκόμαστε σε ένα κόσμο που πιστεύουμε ότι τα συστήματα πρέπει να είναι ισότιμα, συγκρίσιμα. Δεν θέλουμε όμως να ομογενοποιήσουμε την Ευρώπη και τον κόσμο. Από την ποικιλομορφία πρέπει να προκύψει αυτή η σύγκριση και η ισοτιμία και θα πρέπει να υπάρχουν ανάλογες εκπαιδευτικές δομές, θα πρέπει να υπάρχουν ε, ανάλογα συστήματα για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε έναν ανοιχτό και πολυφωνικό χώρο. Αυτά όλα σχετίζονται και με τις επαγγελματικές διαδικασίες και αυτό το θεωρώ θετικό, αλλά είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα δεν τα έχουμε κάνει καλά και δεν τα κάναμε καλά στην εφαρμογή τους. Και ένα από τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε είναι ακριβώς η σχέση με τις εκπαιδευτικέ κοινότητες, με τους καθηγητέ, με την κοινωνία, με του φοιτητέ είπα ότι δεν πρέπει να κάνουμε μόνο για αυτούς, αλλά πρέπει να κάνουμε μαζί με αυτούς. Και μέσω αυτής της διαδικασίας μάθαμε ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε την κοινωνική διάσταση της ε, εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να σχετίσουμε την κατάρτιση μόνο στις ανάγκες της κοινωνίας και της απασχολησιμότητας. Και πρέπει συνεχώς να μαθαίνουμε. Ναι, υπήρξαν σφάλματα, ε, πολλά στην ε, εκτέλεση από κάποιες χώρες, διότι είχαν ως στόχο την ομογενοποίηση των συστημάτων. Κανένας δεν θέλει να ομογενοποιήσει την Ευρώπη. Εμένα δεν μ' αρέσει η ομογενής Ευρώπη. Μ' αρέσει η Ευρώπη της διαφοροποίησης ε, που μπορεί να είναι συγκρίσιμη και συμβατή. Δεν θεωρώ ότι η διαδικασία ήταν αποτυχία, αλλά δεν ε, θεωρώ επίσης ότι ήταν ε, μια διαδικασία μόνο επενδύσιμος. Πρέπει να έχουμε δείκτες, στόχους ε, και από εκεί και πέρα να γίνεται και ένας απολογισμός, διότι η κοινωνία μας ζητά να ενισχύσουμε μεν την παιδεία, αλλά να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Κατανοώ και συμφωνώ, όπως μας είπατε, ε, κάποια πράγματα για την εμπειρία από τη Σλοβενική Προεδρία ότι δεν υπάρχουν αρκετά προσόντα. Ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε διαφοροποιημένη παιδεία και δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι αν δεν έχουμε αυτή την εκπαίδευση με συγκεκριμένες δεξιότητες και προσόντα. Προσπαθούμε λοιπόν να διαφοροποιήσουμε και να κάνουμε πιο ευέλικτη την κατάρτισή μας και μου φαίνεται πολύ λογικό ότι κάποιες χώρες, αναφέρθηκε η Γερμανία, αυξάνουν, τι, αυξάνουν τις ε, επενδύσεις και τα κονδύλια στον προπολογισμό ε, στην έρευνα και στην παιδεία και το μόνο που δεν θα μειωθεί είναι ακριβώς το θέμα της παιδείας. Θα γίνουν ε, περικοπές σε άλλους τομείς, αλλά όχι στην παιδεία. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς αυτή την ε, κατεύθυνση, να υπάρξει ανησυχία για την έλλειψη των κατάλληλων προσόντων, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα νέο προσανατολισμό σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αλλά μέσα σε ένα εξάμεινο προεδρίας είναι λίγο δύσκολο να επισέλθουμε στην αυτονομία πολιτικών αποφάσεων που έχει ε, κάθε χώρα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό όραμα. Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι με την κατάλληλη πολιτική όθηση και με το διάλογο και με την εμπειρία της κάθε χώρας ότι αν δεν επενδύσει δηλαδή στην παιδεία θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια κατάσταση πολύ πιο σοβαρή από αυτήν που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια καλύτερη παιδεία και κατάρτιση. Δεν ξέρω αν είναι για όλους προτεραιότητα, για μένα είναι σίγουρα, για αυτή την Επιτροπή είναι σίγουρα και για την Ευρώπη θα πρέπει να είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Ελπίζω όταν θα συντάξουμε τους προπολογισμού ε, οι ε, πόροι μας να είναι στο ύψος των προσδοκιών μας. Αλλά αν δεν συνεχιστούν οι συζητήσεις, σας διασφαλίζω ότι δεν θα έχουμε τους κατάλληλους πόρους. Ευχαριστώ. Πολύ θαραλέω αυτό το τελευταίο που είπατε και εσείς ε, και οι συναδελφοί σας πρέπει να το θυμούνται. Θα ήθελα κάτι να πω εγώ για τον ανοιχτό συντονισμό. Αυτό είναι η, πόρτα εξόδου από την ε, επικουρικότητα. Οι υπουργοί ξέρουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν άλλο δρόμο, πρέπει να συνεργαστούν. Αλλά επειδή βάζουν πάντα μπροστά την επικουρικότητα, δεν μπορεί κανείς να συνεργαστεί. Και λέμε κάνουμε τον ανοιχτό συντονισμό και από τον ανοιχτό συντονισμό εμάς μας αποκλείουν. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι, αν αποκλείσει τους πολίτες που μέσω ημών παίρνουν μέρο ε, και με την ε, ε, διαδικασία της Μπολόνια, αν, το, αν η διαδικασία της Μπολόνια έχει περάσει από το Κοινοβούλιο, τότε θα είχαν από την αρχή συζητηθεί πολλά προβλήματα από αυτά που υπάρχουν τώρα και θα είχε βρεθεί λύση. Θα είχε τελειώσει το θέμα, θα είχε μπει και η τελευταία λέξη και θα είχαμε προχωρήσει. Εντάξει, τέλο πάντων, α μην θυμώνω πολύ. Ο ανοιχτό συντονισμό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί τουλάχιστον ξέρω ότι είναι κάτι. Αλλά είναι κρίμα που μα αφήνουν απ' έξω από αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό ελπίζω ότι οι κυβερνώντε θα το σκεφτούν αυτό, ότι οι ιδέες που ακούγονται εδώ από την Κομισιόν τα τελευταία πέντε χρόνια και με τη δική μα τη βοήθεια βέβαια, είναι σημαντικές και πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν χρειάζεται να βγει από κάθε ιδέα μας μια οδηγία, αλλά εν πάση περιπτώσει ας είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι. Μιλήσαμε και για κατευθυντήρες γραμμές, ε, δεν θα ήταν ε, κακό να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που ήταν εδώ και βοήθησαν την συνεργασία της ε, Ισπανικής Προεδρίας. Ξέρω ότι είναι πολλά τα προβλήματα που είχατε να αντιμετωπίσετε. Υπάρχει και το θέμα της ε, κρίσης. Ήταν πολλά λοιπόν αυτά που έπρεπε να διαχειριστείτε. Ελπίζω να συνεχίσετε με τη δέσμευσή σας και ελπίζω και η επόμενη Προεδρία να δείξει την ίδια αφοσίωση στα θέματα εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού. Okay. Ah, du bist ja da. Gott sei Dank. Mach's kurz. Ganz kurz. Ich habe schon gehofft, du kommst nicht. So, can we... Uh, we should move to the last item. Πάμε στο τελευταίο σημείο. The last item is the draft... Τελευταίο σημείο, σχέδιο προϋπολογισμού 2011, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Ο κύριος Λόκιγκάρντ είναι ο εισηγητής. Μία σύντομη παρουσίαση να μας κάνει για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Ούτως άλλως το συζητάμε πολύ. Ε, απλώς να πω ότι έχουμε δύο διαδικασίες. Καταρχήν, έχουμε ένα, μία γνωμοδότηση μη νομοθετική, την οποία θα συζητήσουμε. Μία είναι αυτή η ιστορία και την οποία θα ψηφίσουμε. Και παράλληλα με αυτή τη διαδικασία έχουμε και μεμονωμένες τροπολογίες για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής προεπολογισμού Δύο ξεχωριστά πράγματα, τα οποία όμως τρέχουν ταυτόχρονα. Και ε, μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες μέχρι τις 23 Ιουλίου. Ιουλίου. 12 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στις 2 Σεπτέμβρη. Ο κύριος Λόκιγκαρτ έχει το λόγο. Σύντομα και σαφώς και πλήρως παρακαλώ. I'll try to be Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Επιτρέψτε μου να ομιλήσω στην Δανική, διότι το θέμα είναι τεχνικό και είναι πρώτη μου φορά λοιπόν. Μετά την έγκριση της νέας συνθήκης υπάρχει νέα διαδικασία του προϋπολογισμού. Όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο είχε μέχρι τώρα τον τελευταίο λόγο αλλά είναι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθεί κανείς με το Συμβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις για τις διάφορες δαπάνες συνήθως αντιμετωπίζονται μόνο με αιτήματα περικοπών. Εφόσον μάλιστα υπάρχει κρίση, το Συμβούλιο προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα δικαίως μεν. Και έχουν προταθεί περικοπές και για την Επιτροπή μας, για θέματα της Επιτροπής μας. Έχουμε όμως τη συνήθεια να πολεμάμε σκληρά υπέρ των δαπανών μας. Και επομένως να ζητήσουμε τουλάχιστον την επαναφορά στα αρχικά ποσά αν όχι και αύξηση. Τα κράτη-μέλη στις 17 Ιουνίου ενέκριναν αυτή τη στρατηγική του 2020 με πολύ σαφείς στόχους για την παιδεία. Τη στρατηγική αυτή πρέπει να τη σεβαστούμε. Άμα διαβάσετε το σχετικό έγγραφο θα δείτε ότι δεν θεωρείται παρόλα αυτά ακόμη προτεραιότητα. Και δεν προτείνεται καμία αύξηση. τουλάχιστον για ό,τι προβλέπετε για την επόμενη επταετή περίοδο. Αυτό είναι απαράδεκτο, πρέπει να επιμείνουμε τουλάχιστον για την παιδεία. Πρέπει λοιπόν να υποβληθούν προτάσεις, αλλά δυστυχώς για γνωμοδοτήσεις όπως τη δική μου δεν έχω το δικαίωμα να ξεπεράσω τους 1500 χαρακτήρες. Δεν μπορώ να πω λοιπόν όλα όσα θα ήθελα να, να γράψω στη γνωμοδότησή μου. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να στείλω στην Επιτροπή Προπολογισμών ένα σαφέστατο μήνυμα όπου θα τονίζω τη σημασία για μας της παιδείας. Επίσης θα κάνουμε ορισμένες προτάσεις τροποποίησης για τον προϋπολογισμό. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λύγει τον Ιούλιο και ίσως να συνεννοηθούμε πριν από τότε ή τον Αύγουστο με τους Σκιώδης τα θέματα της νεολαίας και της κινητικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικά του χρόνου για τον προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό και γι' αυτό ως Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει και εμείς να επιμείνουμε να μην υπάρξουν αντιφάσεις γιατί αν δεν εγκριθούν επιχορηγήσεις για αυτά τα δύο θέματα δεν ξέρω τι μπορεί να επιτευχθεί. Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν μπορώ να προσθέσω και πολλά. Πρέπει απλώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το Συμβούλιο να μας ακούσει και να δεχτεί τη σημασία της νεολαίας για μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 όλα τα προγράμματα για την νεολαία που έχουμε προβλέψει πρέπει να φροντίσουμε να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Υπάρχουν τα προγράμματα Erasmus Μαρία Κιουρί που είναι πολύ σημαντικά για τους ερευνητές στην Ευρώπη και για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Το Erasmus εξαρτάται για την επιτυχία του από τα πανεπιστήμια μας και άρα χρειάζεται επιγόντως η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και γι' αυτό πρέπει να χορηγηθούν όλα τα κονδύλια τα οποία δικαιούμαστε για τον έρασμο. Όσο για τον University και Business Dialogue και αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως προτεραιότητες. Για το δε πρόγραμμα Μαρία Κιουρί πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες επενδύσεις τουλάχιστον για εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και το ψηφιακό πρόγραμμα. Η επικοινωνία δεν είναι μικρότερη σημασία θέμα και δεν το έχει προσέξει ως έδι η Κομισιόν. Και εδώ πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια. Ξέρω ότι υπάρχει κρίση και ότι θα ζητηθούν περικοπές για τη διοργάνωση σεμιναρίων για δημοσιογράφους. Αυτό θα μπορούσαμε να το δεχτούμε, αλλά και θα καταθέσουμε τροπολογίες και για αυτά. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί ο συντανισμός των δραστηριοτήτων της Κομισιόν ή, ή της Επιτροπής μας. Το λέω και αυτό στη γνωμοδότησή μου, στις Επιτροπής μας μάλλον. Θα δω τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να είναι καλύτερη η πληροφόρηση του πολίτη και του καταναλωτή. Τέλος, τα πιλωτικά ή πειραματικά προγράμματα. Σε λίγο πρόκειται να γίνει μια αξιολόγηση τους από την Κομισιόν και περιμένω με ανυπομονησία να δω τι θα λέει για να συνεργαστώ με τους κοιόδης τους οποίους θα συναντήσω στο Στρασβούργο. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ήβο. Eh, eh, eh, e Από την πλευρά του ΕΛΚ είμαι ο ε, ε, Θα ήθελα να θυμίσω αυτό που περιλαμβάνεται σε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου το Μάρτιο, του Μαρτίου. Μιλούμε για τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011 και εκεί είχαμε αναφέρει τις δράσεις για τους νέους ανθρώπους. Είναι πολυετή προγράμματα αυτά, όπως ας πούμε οι νέοι σε δράση, πολιτιστικά προγράμματα, η, η ε, για παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι Special Olympics, η Ευρώπη των πολιτών. Στο σχέδιο του προπολογισμού αναφέρονται ε, κάποια αριθμητικά στοιχεία. Ε, μιλούμε δηλαδή για 28 εκατομμύρια. Το Κοινοβούλιο είπε ότι αυτά τα προγράμματα είναι απο, αποκλειστική προτεραιότητα και αυτό προκύπτει και από το ψήφισμα του Μαρτίου. Το ξαναλέω. Ο προπολογισμό είναι περιορισμένος. Και σας παραπέμπω και στο έγγραφο του κυρίου συζητητή. Ε, δεν μπορώ τώρα να διαβάσω το, το επίθετο, είναι λίγο δύσκολο. Λέει εδώ στο κείμενο ότι παρά της ε, ε, εφαρμογής που ξεκινάει από τον τίτλο 14 για την διαβιομάθηση, πρέπει να έχουμε μια, ένα επίπεδο εφαρμογής που θα πρέπει να φτάνει στο 100% που είναι πολύ υψηλό. Ο, το σχέδιο προπολογισμού του 2011 αυξάνει τι ε, δεσμεύσει και είναι πολύ περιορισμένο. Δηλαδή αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, να το έχουμε υπόψη, γιατί αυτά τα σχόλια τα είχε κάνει τότε ο ε, εισηγητή. Και αυτό είναι που είχε αναφέρει και τα βασικά, τις βασικές άγουσες αυτής της ε, γνωμοδότησης. Άλλο ένα, άλλη μια παρατήρηση. Εδώ μιλούμε για τις αρμοδιότητες, για τον αθλητισμό. Πολλά μέλη αυτής της α, α, πολιτικής ασχολούνται και με τον αθλητισμό. Ξεκινά το πρώτο πρόγραμμα για τον αθλητισμό το 2012 και τι γίνεται για, αυτό το, για αυτές τις παρασκευαστικές ε, διαδικασίες για το πρόγραμμα αυτό. Ο, ο, προϋπολογισμός από 3 εκατομμύρια γίνεται ένα. Ε, και πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό. Η, αυξάνουμε και προσθέτουμε συνέχεια προγράμματα και μειώνουμε τους σπόρους. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Και μια άλλη ερώτηση που ίσως να είναι σημαντική όταν μιλούμε για την Europol. Κύριε Λόκιγκαρντ, ξέρετε πόσο, σημαντική, πόσο σημαντικό είναι το ερώτημα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα το θέμα της Europol. Μιλούμε, τα, τα ΜΜΕ λένε για 6, έλεγαν για 6 εκατομμύρια, τώρα είχαν πάει στα 5. Ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερες προσπάθειες για να βελτιώσουμε το τι βγαίνει από τα ΜΜΕ. Οπότε θα ήθελα αυτό να το λάβετε υπόψη σας με κάποιο τρόπο στην έκθεση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κανένα τον λόγο, να κάνω και εγώ δύο παρατηρήσει. Κύριε Λόκεγκαρτ, δεν υπάρχει ε, καμία γραμμή για τον, στον προπλογισμό για, τις, ε, για τους νέους σε κίνηση. Αυτό υπάρχει στην διαβιομάθηση, υπάρχει στην, στους, στην νεολαία σε, έτσι γενικά, αλλά ως γραμμή για, ε, συγκεκριμένα για το νέο σε δράση Δεν υπάρχει. Καλό είναι αυτό γιατί μπορούμε έτσι να προωθήσουμε καλύτερα τα προγράμματά μας εκπαίδευση. Ε, για τον αθλητισμό εντάξει είναι γελία η κατάσταση, ναι. πολύ λιγότεροι οι πόροι, έχουμε ε, προσθέσει προγράμματα, ε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι με τις δράσεις που θέλουμε να προωθήσουμε. Και όντω νομίζω ότι πρέπει και να δούμε την κατάσταση με τα ΜΜΕ. Το θέμα δεν είναι πόσα θα δώσουμε στα, ε, σε εκστρατείες ε, ενημέρωσης κτλ ή τι θα λένε τα, τα ΜΜΕ. Το θέμα δεν είναι να δώσουμε περισσότερα χρήματα, είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα. Το ίντερνετ υπάρχει, τα ΜΜΕ υπάρχει, πρέπει να φτάσει το μήνυμά μα στου πολίτε με κάποιο τρόπο. Εκεί πρέπει να βελτιωθούμε. Αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα περισσότερα χρήματα. Η συντόνια Ελιζαμπέτα είναι μια εξαιρετική συνάδελφος η οποία έχει αναλάβει την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να, την, να της δώσουμε έτσι κι άλλη τροφή για σκέψη για να μπορέσει να συμπληρώσει την ε, γνωμοδότησή της. Εμείς έχουμε προγράμματα τα οποία ούτως ή άλλως τρέχουν. Βρίσκονται να εξελίξει 7 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα κόψουμε ξαφνικά. Δεν βλέπω δηλαδή στον τομέα ε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε μάλλον τα προγράμματα ξαφνικά ή να αναβάλουμε. Εντάξει, αν δούμε ότι κάποιο ε, πρόγραμμα σε κάποιο τομέα δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει απορροφηθεί όσο πρέπει, ίσω να πρέπει όντω να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο τρόπο, να βελτιώσουμε το πρόγραμμα, να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Εκεί ναι, στην παιδεία το κάνουμε, στου νέου το κάνουμε, στου πολίτε επίση. Οπότε εγώ συμφωνώ με τον, ε, με τον ε, Ήβο. Γιατί έχουμε, πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τι εταιρικέ σχέσει, τη συμπράξη των πόλεων. Έχουμε που παλεύουμε για το θέμα αυτό τόσα χρόνια. Και το θέμα της, ε, το European Citizenship νομίζω ότι δεν το έχει αναλάβει, δεν είναι στις αρμοδιότητες της κυρίας Βασιλείου. Ε, δεν ξέρω ποιος, αν θέλει ο, ε, ο εισηγητής να κάνει κάποιο σχόλιο, η Κομισιόν θέλει, ναι. Η Κομισιόν θέλει το λόγο. Okay. <laughs> Α, ναι. Λοιπόν, πολύ σύντομο θα είμαι. Υπάρχουν προγράμματα όπως η επικοινωνία και θέματα ηθαγενείας που δεν είναι της δικαιοδοσίας μας για τον αθλητισμό που αναφέρθηκε συχνά. Άμα δείτε τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό της Κομισιόν, ο αθλητισμός είναι ο μόνος τομέας όπου η Κομισιόν έχει ήδη προβλέψει κονδύλια για το 2011 στον προϋπολογισμό. Τα άλλα παραμένουν εκκρεμή για τις δύο αρχές του προϋπολογισμού. Αυτό δείχνει ότι η Κομισιόν είναι υπέρ της δαπάνησης αυτών των χρημάτων για τον αθλητισμό και πάνω από το 1 εκατομμύριο. Και πέρυσι είχαμε προβλέψει ένα ποσό το οποίο αύξησε τελικά το Κοινοβούλιο. Απάντως δείχνει ότι δεν είμαστε κατά. Ακριβώς για την προετοιμασία του αθλητικού προγράμματος 12-13. Κύριος Φύσας, τελευταίος. Ναι, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα του αθλητισμού. Φοβάμαι ότι δεν είναι πολύ σαφή η σημασία που του δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη σημασία μάλλον τη δίνει το Κοινοβούλιο και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εμείς καταφέραμε να αυξηθεί ο προπολογισμό το να ξεκινούμε από τόσο χαμηλή βάση από αυτήν που έχουμε, όταν ε, μάλιστα υπάρχουν και νέε αρμοδιότητε που προκύπτουν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ε, με οδηγεί στην κατάληξη ότι μιλάμε για γελία πράγματα. Υπάρχει ένα ποσό, αλλά δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο που θα πρέπει να κάνει προσπάθειες για να αυξηθεί αυτό το ποσό. Το ποσό. Θα το κάνουμε, σίγουρα θα το κάνουμε, αλλά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμό, ε, τι νέε δικαιοδοσίε υπάρχουν σε θέματα αθλητισμού και να παρουσιάσει ένα σχέδιο το οποίο θα είναι αξιοπρεπές και επαρκές για τους νέες φιλοδοξίες που υπάρχουν σε θέματα αθλητισμού. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, κλείνουμε τη συζήτηση να σας πω ότι Έχουμε συλλέξει κάποιες δράσει. τις έχουμε υποβάλει για να, μας ε, για να κάνει παρατηρήσεις της Κομισιόν, αλλά αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσει θα πρέπει να υποβληθούν επισήμως ω τροπολογίε στη, στην ε, γνωμοδότηση του κυρίου Λόκεγκαρτ. Ω τροπολογίε. Όχι ω σκέψει, γιατί οι σκέψει έχουμε μπόλικε. Απλώς για να δούμε και ποιε είναι οι παρατηρήσει τη Κομισιόν. Είδα και στην ε, Νέα Αφρική τι γίνεται με τα παιδιά και με τι μπορούν να κάνουν με το ποδόσφαιρο που παίζουν στο δρόμο. Πραγματικά είναι κάτι εκπληκτικό. Ίσως ε, θα μπορούσαμε κάτι παρόμοιο να κάνουμε και εμείς εδώ και το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, όλα όσα έχετε υποβάλει ως πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να επαναυποβληθούν ως τροπολογίες. 23 Ιουλίου σας είπα ότι είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Και τον Σεπτέμβρη ξεκούραστη, θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ που βοηθήσατε και δεν δαπανίσαμε πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστώ η Πρόεδρος και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Καλό σας απόγευμα. Α, όχι, η κυρία Χάνιμπαλ θέλει κάτι, παρακαλώ. Συγγνώμη, Πρόεδρε, ξέρω ότι όλοι θέλουμε να φύγουμε, αλλά έχω κάποια σχόλια για, τους, για τις αποφάσεις των εισηγητών. Των συντονιστών, συγγνώμη. Για το σημείο 3, και την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Εκπαιδευτική Κατάρτιση και την, εκπαιδευτική... και την ε, Εκπαίδευση. Ε, μήπως θα μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό το κομμάτι στα πρακτικά για την επαγγελματική κατάρτιση, συγγνώμη. Ε, επίσης, σημείο 3. Για, την, για τις νέες γνωμοδοτήσεις ίδιας πρωτοβουλίας. Η δεύτερη ο ρόλος των νέων μέσων ε, και της νέας εξωτερικής πολιτικής ε, και των νέων μέσων πολιτισμού. Εγώ ε, το έχω ξαναφήξει το θέμα αυτό, αλλά από ό,τι κατάλαβα και οι συνάδελφοί μου συμφωνούν ότι εσείς θα το αναλάβετε ως πρόεδρος και μέλος του ΕΛΚ. Και τώρα λέει ότι θα το πάρει η Άλντε την έκθεση αυτή. Και δεν θεωρήσαμε ότι αυτό είχαν αποφασίσει οι συντονιστές. Λοιπόν, το πρώτο είναι λάθος, θα γίνει, το δεύτερο είναι σωστό. Εγώ είδα το αίτημα της Άλντε και χάρηκα που το υπέβαλαν. Αν δεν το υπέβαλαν θα το έπρεπε να το αναλάβω εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ που θέλω να κάνω αυτή την έκθεση. Εγώ ως ε, πρόεδρος δεν θέλω να, να, λαμβάνω τα πάντα, θέλω να αφήνω χώρο και στους ε, συναδέλφους. Είχα λοιπόν αυτή την ιδέα. Χτε το βράδυ έκανα μια στρογγυλή τράπεζα γιατί θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή να μιλήσουμε για την διάρθρωση τη υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Αν δεν μιλήσουμε τώρα για τον πολιτισμό στι εξωτερικέ υποθέσει, πότε θα το κάνουμε, όταν θα έχουν δημιουργηθεί όλα και θα μα έχουν ξεχάσει. Γι' αυτό χάρηκα που το πρότεινε η Άλντε. Και είπα επιπλέον, η Άλντε δεν ήταν η σειρά τη, α πούμε. Κάποιο άλλο θα έπρεπε να το έχει πάρει, θα ήθελα να το έχει πάρει. Η Άλντε όμω, αφού το υπέβαλε, δεν μπορούσα να του πω εγώ, Όχι, δεν θα το αναλάβετε, το αναλαμβάνω εγώ. Πρέπει όμω να είμαστε προσεκτικοί. Επειδή η κυρία Σάλκη έκανε την πρόταση αυτή, εγώ τη το ανέθεσα και, είπε ότι, και είπαμε ότι φυσικά είναι σημαντική η γνωμοδότηση και είπα πολύ συγκεκριμένα ότι φτάνει πλέον με του φιλελεύθερου. Έχουν λάβει πολλά, έχουν αναλάβει πολλέ. ίσως μετά να αναλάβει η Γκουε ή άλλες ε, πολιτικές ομάδες. Το είπα σαφέστατα ότι φτάνει με τους ε, ε, φιλελεύθερους, έχουν αναλάβει πολλά και το δέχτηκαν. Έκαναν όμως το αίτημά τους, δέχτηκαν να αναλάβουν την γνωμοδότηση. Αυτά. Με την τροποποίηση λοιπόν που ζητάτε να γίνει για το σημείο 2, θα το διορθώσουμε, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε οι συντονιστέ, εντάξει, γίνονται δεκτέ αποφάσει. Πολύ ωραία. Διάφορα δεν υπάρχουν, ε, τα έχουμε συζητήσει όλα. Παρακαλώ, έχετε κάτι στα διάφορα. Για να διευκολύνουμε λιγάκι την επόμενη συνεδρίαση, Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε και το απόγευμα της Τετάρτης για την επόμενη συνεδρίαση. Εντάξει, μπορούμε να το δούμε, δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε τώρα. Απλώς το λέω. Ε, θα δούμε. Δεν συνεδριάζουμε για να συνεδριάζουμε. Αν ε, χρειάζεται το απόγευμα, θα χρησιμοποιήσουμε και το απόγευμα, φυσικά. Μπορούμε να το δούμε όμως. Ε, εντάξει, να προσπαθήσουμε δηλαδή να είναι ε, αυστηρή, αυστηρό το χρονοδιάγραμμά μας για να τελειώσουμε νωρί. 13 Ιουλίου η επόμενη συνεδρίαση, 14 Ιουλίου επίση. Ίσως με το απόγευμα, ίσω χωρί το απόγευμα. Μέχρι τότε Καλό σας απόγευμα και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστή η πρόεδρος της και εμείς. Καλό σας απόγευμα.